colleagues, I Λοιπόν, συνάδελφοι, βλέπω ότι αδειμονείτε να ξεκινήσουμε. Χαιρόμαστε που έχουμε ανάμεσά μας την Επίτροπο Κούνεβα, η οποία συχνά έρχεται να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις ε, που έχουν οι στην Επιτροπή και χαίρομαι που σήμερα θα μας παρουσιάσει τον ε, πίνακα του 2009 πίνακα επιδόσεων και θα δούμε κατά πόσον αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν τον πίνακα επιδόσεων και χαιρόμαστε που για πολλά χρόνια στην Επιτροπή μας ασχολούμαστε με τα αποτελέσματα του πίνακα για την αγορά Θέλαμε λοιπόν να δημιουργηθεί αυτός ο πίνακας επιδόσεων για να έχουμε κάποια στοιχεία μετρήσιμα για τα αποτελέσματα. Χαιρόμαστε λοιπόν που η πρωτοβουλία αυτή έχει προθεθεί και έχει προθεθεί με τον γνωστό ενθουσιασμό της κυρίας Κουνέβα. Παρακαλώ και το λόγο και μετά θα ακούσουμε τις ε, ερωτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι απόλυτα αληθές ε, και δεν υπερβάλλω εάν ε, αναφέρω πως αυτός ο πίνακας επιδόσεων έχει εμπνευστεί από το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση, είναι πολύ καλύτερη θα λέγαμε από την πρώτη εκδοχή του και χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω το δεύτερο πίνακα δώσουν για τον καταναλωτή. Ο πρώτος πίνακας ε, ήταν αποτέλεσμα μετά πολλών συζητήσεων στην Επιτροπή σας. Εξαιτήμη ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σας και την υποστήριξή σας αλλά και την οικονομική επίσης υποστήριξη που χορηγήσατε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα 2008 αλλά και 2009. Χωρίς λοιπόν αυτή την απτή υποστήριξη θα είχε καταστεί δυνατόν να έχουμε στα χέρια μας αυτό το πίνακα επιδόσεων. Αλλά πρωτού να παρουσιάσω τα αποτελέσματα του δεύτερου πίνακα, να σα υπενθυμίσω για ποιο λόγο αυτή η πρωτοβουλία είναι τόσο σημαντική. Διότι από τότε που φασίσαμε την ύπαρξή του έχουν, έχουν γίνει νέες εξελίξεις και Αναφέρομαι στην οικονομική κρίση, αλλά αν θέλουμε πολιτικές οι οποίες θα αποδίδουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τον καταναλωτή, θα πρέπει να είμαστε πιο ε, υπεύθυνοι και να κατανοήσουμε καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Εδώ, του λοιπόν, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία για να δούμε πώς λειτουργούν οι αγορές και πώς ε, ε αντιδρούν οι πολίτες, οι καταναλωτές. Οι πίνακες αυτές ε, μετράνε την, κατα, την ικανοποίηση του καταναλωτή, τις τιμές που καταβάλουν και τις ε, δυνατότητες που τους δίνουν. Παρατηρούμε επίσης τις αγορές από την πλευρά του καταναλωτή και νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, το γνωρίζετε. Ότι δηλαδή βλέπουμε τις αγορές από την πλευρά του καταναλωτή και από την πλευρά της ε, αποτελεσματικότητας. και θα λέγαμε ότι είναι πιο αποτελεσματική πρακτική που έχουμε ακολουθήσει. Να αναφερθώ τώρα στην πρόσφατη εκδοχή του πίνακα. Όπω γνωρίζουμε είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται και τα στοιχεία που έχουμε διαθέσει μα είναι ατελή. Πολλά έχουν να γίνουν ακόμα προκειμένου να έχουμε, την απαραίτητη διαφάνεια στις αγορές μας και να επιτραπεί απόλυτη εποπτεία των μεγαλύτερων αγορών. Η δεύτερη εκδοχή λοιπόν του πίνακα ε, έχει αποφέρει κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Θα ξεκινήσω με τα σκάλες ειδήσει. Το πιο θετικό αποτέλεσμα είναι πως ε, παραδοσιακά ο τομέας μόνο των παραδοσιακών αγαθών ε, συμπεριφέρεται αρκετά ικανοποιητικά. Αναλύθηκαν 19 τομείς των καταναλωτών είπαν ότι είναι ικανοποιημένοι με τα αγαθά τα οποία αγόρασαν αλλά και από τα καταστήματα τα οποία αγόρασαν τα αγαθά αυτά. Καλύψαμε λοιπόν πάρα πολλά αγαθά όπως ε, τα κρατικά, τα οχήματα, τις ε, νέες τεχνολογίες, ε, ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισμό και βιβλία. Ε αγορές των αγαθών αυτών συνήθως συμπεριφέρονται καλύτερα από ότι οι αγορές ε, των υπηρεσιών. Αλλά κλάδοι όπως οι ασφάλειες και οι τηλεπικοινωνίες ε, σύμφωνα με δύο στους καταναλωτές ε, είναι ικανοποιητικές και μόνο 11% των καταναλωτών ανέφεραν προβλήματα με αυτές τις δύο υπηρεσίες. Επίσης ήταν εύκολο να κάνουμε σύγκρισης. και στον τομέα των ασφαλείων όπου παρατηρήσαμε ότι ένας στους τέσσερις ε, καταναλωτές άλλαξε ασφάλεια στο όχημά του. Ε, το τομέα των τηλεπικοινωνιών επίσης θα πήγε αρκετά καλά, ειδικά σε ό,τι φορά την αλλαγή παρόχου. 22% των καταναλωτών άλλαξαν τον πάροχο στο ίντερνετ παρά το ότι πολλοί καταναλωτές αναφέρουν προβλήματα για την αλλαγή παρόχου. Η τιμή για την αλλαγή παρόχου είναι ιδιαίτερα υψηλή για, στον τομέα των κινητών τηλεφώνων και 67% των καναλωτών μπόρεσαν να ε, κάνουν μια αποτελεσματική σύγκριση και να τροποποιήσουν, να αλλάξουν τον, τον πάροχο. Αυτό είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό, το υψηλότερο θα λέγαμε της έρευνας. Θα μου πείτε γιατί ε, εστιάζω στο ζήτημα του κόστους της αλλαγής παρόχου. Διότι οι καταναλωτές, μάλλον η για τους καταναλωτές αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η, από ό,τι παρατηρήσαμε, ο ανταγωνισμός λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος του καταναλωτή. Λοιπόν, η διευκόλυνση της ε, αλλαγής ε, παρόχου σε αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες. Τώρα, τα στοιχεία που έχουμε για τους καταναλωτές δείχνουν ότι οι τάσεις είναι πολύ ικανοποιητικέ. Η συμμόρφωση με την ε, νομοθεσία ήταν ένα από τα ερωτήματα, το πώς προστατεύονται οι καταναλωτές από τα ισχύοντα μέτρα και πώς εύκολα μπορούν να τύχουν επανόρθωση. Είδαμε από τη χώρες όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Ολλανδία τα πήγαν πολύ καλά σε σχεδόν όλους τους δείκτες. Και είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι μια σειρά νέων κρατών όπως Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Λετωνία και Εστονία καταγράφουν σημαντική πρόοδο σε όλους τους δείκτες. Και τώρα να αναφερθώ και στα λιγότερο καλά νέα. Ε, όταν ε, τα πράγματα δυσκολεύουν, ορισμένες ε, υπηρεσίες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά και προς όφελος του καταναλωτή αυτό αυτή είναι η κλάδη της ενέργειας, ο τραπεζικός κλάδος και οι συνδρομικές και οδικές μεταφορές το 1 τρίτο των καταναλωτών είναι ικανοποιημένοι από την παροχή ενέργειας εδώ. Είναι ένα στο μέσο που 3 στους πέντε καταναλωτές αναφέρουν αύξηση τιμών. αλλά και χαμηλή ικανοποίηση. Ο τομέας ενέργειας είναι ένας κλάδος όπου δύσκολα κανείς μπορεί να αλλάξει πάροχο. Λιγότερο από 10% των καταναλωτών άλλαξαν πάροχο τα τελευταία δύο χρόνια στον τομέα του αερίου ή του πετρελαίου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από τους φόρους, ο ελεκτρισμός των Γερμανία και το Βέλγιο είναι 5% υψηλότερο το κόστος από ό,τι στην Πολωνία οι τραπεζικές εργασίες και εδώ είναι πιο υψηλές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει χαμηλό ποσοστό αλλαγής παρόχου. Κατά μέσον όρων μόνο 9% των χρηστών αλλάζουν τράπεζες και 24% των καναλωτών θεώρησαν ότι είναι δύσκολο να μπορέσουν να συγκρίνουν τις ε, προσφορές που κάνουν οι πάροχοι. Επίσης, ε, πολλές προφορίες αποκρύβονται από τους καταναλωτές. Να κάνω ένα παράδειγμα. Το, στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν ότι οι τράπεζες κερδίζουν από τις προμήθειες τις οποίες δεν γνωρίζουν καν τις περισσότερες φορές οι καταναλωτές. Βρήκαν ότι 20% των καταναλωτών δεν εγνώριζαν για τις ε, προμήθειες που πρέπει να πληρώνουν σε περίπτωση που ο λογαριασμός τους ε, στο, ε, παραμείνει ακάλυπτος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Πρέπει επίσης να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ε, υπηρεσίε που παρέχουν οι τράπεζες, ειδικά στην περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης. Τέλος, να αναφέρω τις οδικές και τις ηρωνικές μεταφορές που και αυτές προκαλούν πρόβλημα. Η ικανοποίηση σε τον κλάδο είναι ιδιαίτερα χαμηλή και όχι μόνο για την τιμολόγηση αλλά και για την προσφορά υπηρεσιών. Ε, οι αστικές υπηρεσίες θεωρούνται ότι είναι ιδιαίτερα ακριβείς και οι θεωρούν ότι οι εταιρείε δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για τους επιβάτες. Όταν μιλάμε για την αρχή τώρα της επικουρικότητας ό,τι αφορά τις ε, αστικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για όλους όσους ε, καταρτίζουν και χαράσουν τις πολιτικές αποφάσεις λοιπόν, όπως και μετά από το δεύτερο πίνακα επιδόσεων. Να, εδώ ανοίγω μια παρένθεση να σας πω ότι από τον Μάρτιο 2009 θα σας παρουσιάσω την πρώτη συνέχεια που δώσαμε μετά από τον πρώτο πίνακα επιδόσεων και θα είμαι έτοιμη λοιπόν, αν φυσικά με προσκαλέσετε, να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διότι αυτός θα είναι ένας κλάδος που θα πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ε, σύμφωνα με την κατάργηση των εμποδιών και των φραγμών. Θα σας αναφέρω λοιπόν τα συμπεράσουμε μετά από τον πρώτο πίνακα. Τώρα, το δεύτερο βήμα ποιο είναι. Θα θέλω να εστιάσω στον τομέα της ενέργειας και του ηλεκτρισμού για το 2009. Αυτό φυσικά θα το κάνουμε από κοινού με τον Επίτροπο Πίλμπαξ. Θα καταρτήσουμε έκθεση για να εξετάσουμε πώς λειτουργεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές Κανοντά την συγκρισιμότητα των προσφορών, την τιμολόγηση και τις εμπορικέ πρακτικέ. Επίση, ε, περιμένουν να σημαντική ε, βοήθεια από το Φόρουμ των Πολιτών που θα εξεχθεί για δεύτερη φορά τον Οκτώβριο, πρώτη φορά διεξήχθη πέρυσι, για ανάλυση των ε, συνθήκων θα συμβάλλει σημαντικά για την ίσχυση τη θέση των οργανωτών και να μπορούν να κάνουν σωστέ επιλογέ και να δραματίσουν ρόλο σε μια σωστά λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Θα ενδεχόμενοι τώρα στι προτάσει σα και την εξωτερική έκθεση τη κυρία Χατ από πέρυσι, όπου τονίσατε πως ε, αυτό ο πίνακα επιδόσεων θα πρέπει να γίνει πιο προσβάσιμο και ανοιχτό στο ευρύτερο κοινό και να δημιουργηθεί καλύτερη επίγνωση να μεταφραστεί φυσικά σε όλες τις ε, γλώσσες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα και τις ε, συστάσεις και Επίσης τονίσατε πως η σημασία της ταινής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη και πολύ σωστά το πράξατε θα βοηθήσει στο να βελτιώσει τα πληροφορίες μας. Χρειάζεται λοιπόν συμμετοχή των εμπλεκομένων, των φορέων κλπ. Έχουμε, πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις ε, στατιστικές αρχές και τις οργανώσεις των καταναλωτών. Τέλος, ε, μιλήσω στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο ήδη ανέφερα. Απέφυγα να αναφέρω τις εξελίξεις στο διασυνοριακό εμπόριο, διότι πρόκειται να ε, κυκλοφορήσουν εκθέσεις ε, περί αυτού συντόμως. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για μια σφαιρικότερη έκθεση για την γεωγραφική κατανομή, καταμερισμό της ε, λιανικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προτίθεμεθα να συντάξουμε τον Ιούνιο. Αυτό λοιπόν θα είναι μια συντονισμένη προσπάθεια, τονίζω λοιπόν ότι είναι συντονισμένη προσπάθεια ε, όλων των επιτρόπων που ασχολούνται με θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι πραγμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε διασυνοριακό επίπεδο. Έφτασε η ώρα λοιπόν η Επιτροπή να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών για την ιστορική αγορά, για, την ε, online, ε, για το online γενικό εμπόριο. Ελπίζω να μπορώ να βασιστώ σε εσά προκειμένου να να δημιουργήσουμε αποτελεσματικότερα λειτουργούσες ε, αγορές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υποστήριξη που μου μέχρι τώρα και Περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Τις ερωτήσεις, ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο της εισήγησης και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και μελλοντική εργασία σε σχέση με τις αγορές ενέργειας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε ερωτήσεις. Εγώ θα περιμένω στο τέλος μέχρι να ακούσω τα άλλα μέλη. Λοιπόν, η κυρία Χέτ καταρχήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, Πρόεδρε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Κούνεβα για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση αυτή ε, χάρηκα ιδιαίτερα, ιδιαίτερα όταν άκουσα τα θετικά σημεία που θίξατε, αλλά βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αρνητικές πτυχές και αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και τι να καταφέρουμε καλύτερα. Χαιρόμαστε λοιπόν για αυτό τον απολογισμό θετικό ή αρνητικό και χαιρόμαστε διότι ο πίνακας επιδόσεων είναι διαθέσιμο σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές κοινοτικές γλώσσες και θα είναι διαθέσιμος και στο διαδίκτυο για τις ενώσεις καταναλωτών, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να δουν τα αποτελέσματα οι ίδιοι. Ένα ερώτημα που θα ήθελα να υποβάλω αφορά το σύστημα ταξινόμησης. Θα πρέπει να έχουμε συγκρίσιμα συστήματα ταξινόμησης για να μπορούμε να κρίνουμε εισάξια. Δηλαδή, ως προς τις προσφυγές θα πρέπει να έχουμε μία σωστή εκτίμηση, άρα μία ίση βάση εκτίμησης. Ίσως αυτό είναι δύσκολο, αλλά σε λίγα χρόνια ίσως μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή τη βάση εκτίμησης. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του πίνακα επιδόσεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάιλερ. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, κυρία Επίτροπε, διότι εργαζόσαστε πολύ σκληρά για το ζήτημα αυτό. Είχαμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων και ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο σας υποστηρίζει. Άκουσα, μάλλον διάβασα το γερμανικό τύπο πριν έρθετε εδώ επί του θέματος και φαίνεται ότι υπάρχει μία καλή ε, διανομή και τεκμηρίωση. μετά από το πρώτο ευρωβαρόμετρο και το σχετικό σοκ, κάτι έκανε το Κοινοβούλιο το οποίο υποβοήθησε την κατάσταση. Όταν αλλάζει κανείς πάροχο, αυτό δεν είναι αφεαυτού ένας στόχος, αυτός σκοπός δηλαδή. Θα πρέπει να σχετίζεται με βελτιώσεις για τον καταναλωτή και επίσης μία κίνηση στην αγορά. Κάτι το οποίο διαπιστώνουμε στη γερμανική αγορά για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνιση. Δεν υπάρχει θέμα τιμολογίων μόνο, αλλά και θέμα ποιότητας. Και μιλάμε φυσικά και για διαφάνεια. Λοιπόν, ως προς τον τομέα της ενέργειας έχω ορισμένες ερωτήσεις. Είπατε ότι μελλοντικά θέλετε να ε, ασχοληθείτε περισσότερο με αυτό. Εγώ όταν άλλαξα σπίτι, άλλαξα και πάροχο και είδα ότι αυτό είναι πολύ εύκολο, τουλάχιστον στη Γερμανία. Πολλοί Γερμανοί, μερικοί Γερμανοί βεβαίως είναι επιφυλακτικοί γιατί θεωρούν ότι θα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για αλλαγή φορέα ή παρόχου. Μπορεί πραγματικότητα να μην το αντικατοπτρίζει αυτό, αλλά δεν το ξέρει ο καταναλωτής. Γι' αυτό χρειάζεται η διαφάνεια. Σε ορισμένα κράτη-μέλη η διαφάνεια αυτή δεν ήταν αναπόσπαστο τμήμα του πακέτου όπως στην Σκανδιναβία όπου τα πράγματα είναι πιο ανοιχτά. Άρα θα σας υποστηρίξουμε στην αγορά ενέργειας. Αναφερθήκατε σε ορισμένα κριτήρια δηλαδή εμπορικές ε, πρακτικές, αλλά θα ήθελα να λάβετε υπόψη και ένα άλλο σημείο, δηλαδή τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Παρατήρησα στη γερμανική αγορά ότι υπάρχουν ε, ορισμένοι παραδοσιακοί πάροχοι ενέργειας όπου ε, προβαίνουν σε τιμολογήσεις ε, πηγών ενέργειας που είναι φιλικές προς το χρήστη και αφορούν ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας και όχι πυρηνικά, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και αυτό βεβαίως σχετίζεται με τις παραπλανητικές διαφημίσεις που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος ε, Μάντερς. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, κυρία Επίτροπε. Ήταν πολύ θετική η παρουσίαση αυτή και υποστηρίζω και την ιδέα ότι θα πρέπει να ικανοποιήσουμε τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την αγορά ενέργειας, νομίζω ότι δεν υπάρχει ακόμα εσωτερική αγορά για την ενέργεια. Αναφερθήκατε στη ε, Γερμανία και την Ολλανδία, δηλαδή πριν από τη φορολόγηση έχουμε να κάνουμε με μια τιμή η οποία διπλασιάζεται στη συνέχεια. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε άλλες χώρες και δεν μπορούμε πολλές φορές να παραγγείλουμε ε, ενέργεια μέσω διαδικτύου. Επίσης μπορεί κανείς να αλλάζει πάροχο αλλά μπορεί ε, πρέπει να λάβει την ενέργεια από την ίδια αγορά. Άρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, άρα οι τιμές είναι οι ίδιες. Ως προς την αλλαγή παρόχου ενέργειας δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ελπίζω να σας, να σας υποστηρίξει ο κύριος Πι έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια εσωτερική αγορά ενέργειας την επόμενη θητεία, έτσι ώστε ο τελικός χρήστης να μπορεί να ε, λαμβάνει ενέργεια από που θέλει με βάση ενιαίες τιμές και μέσω διαδικτύου. Μιλάτε για την ικανοποίηση των ε, καταναλωτών. Δεν υπάρχει υποστήριξη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και από τη χώρα μου, από την Ολλανδία. Αν ρωτήσετε τον καταναλωτή κατά πόσο είναι ικανοποιημένος με το προϊόν στην εσωτερική αγορά, είναι μεν ικανοποιημένος. Αν όμως τους ρωτάτε τι θέλετε από την Ευρώπη, λένε δεν θέλουμε άλλη Ευρώπη. Πώς μπορούμε να χτίσουμε μία γέφυρα για να υπάρχει υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ισχύει για την αγορά προϊόντων. Άλλη μία υπόδειξη. Πολλές φορές ε, μιλάμε, ρωτάμε κατά πόσο υπάρχει ικανοποίηση από την αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων και την ε, κατάσταση της αγοράς. Ίσως θα μπορούσατε να έχετε ένα κουτί υποδείξεων και παραπώνων μέσω διαδικτύου και να ζητάτε γνώμες μέσω ιστοτόπων από τους καταναλωτές πώς μπορεί να επιληθεί η χρηματοπιστωτική κρίση έθνης. Μπορεί ένας μέσα στα εκατομμύρια να δώσει μια λύση την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σε πολλές επιχειρήσεις όταν φεύγει κανείς από την επιχείρηση υπάρχει ένα κουτί που μπορεί κανείς να ρίξει τις ένα χαρτί με τις υποδείξεις του. Το έχουμε και κάτω στην καντίνα μας. Άρα οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν υποδείξεις για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές, έτσι ώστε να εργαστούμε θετικά. και να επεκτείνουμε αυτή την υποστήριξη για την Ευρώπη από όλους γενικά. Χωρίς μικρόφωνο η Πρόεδρος. η, Επίτροπος. Σας ευχαριστώ. Θα αρχίσω με την ταξινόμηση των καταγγελιών. Είναι πολύ σημαντικό. Κάτι που λείπει σε όλη την Ευρώπη για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές και χωρίς να υπάρχει κοινή βάση για ταξινόμηση των καταγγελιών δεν μπορούμε να δώσουμε και αυτή την αίσθηση της ενότητας. Και η Federal Trade Commission για παράδειγμα στις Ηνωμένε Πολιτείε, που ε, είναι ισχυροί γιατί υπαγορεύουν και την πολιτική διότι οι καταγγελίες των καταναλωτών δεν καταλήγουν μόνον στον Ombudsman ο οποίος εγκύπτει στη συγκεκριμένη καταγγελία και ενδεχομένω να ικανοποιηθεί ο συγκεκριμένο καταναλωτή, αλλά οι καταγγελίε αυτέ μαζεύονται αν είναι πολλέ, α πούμε για τι τηλεπικοινωνίε ή για την ενέργεια ή για ε, ε, πλαστά προϊόντα κ.ο.κ. Αυτό αρχίζει πια και υπαγορεύει την πολιτική. Δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την πολιτική που ασκείται στο συγκεκριμένο τομέα. Αν δείτε στην ανακοίνωση στην σελίδα 6 αναφέρομαι σε αυτό ακριβώς το θέμα. Αυτές τα παράπονα ή καταγγελίες των ε, καταναλωτών είναι βασικός δείκτης. Συλλέγονται τώρα από τις εθνικές αρχές της χώρες μέλη, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν εναρμονιστεί οι διαδικασίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν επιτρέπουν έτσι να γίνει σύγκριση μεταξύ αγορών και χωρών. Έγινε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για την ταξινόμηση των ε, καταγγελιών των καταναλωτών και ε, τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν τέτοια ιδέα. Βέβαια δεν θα περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες βιομηχανίες. Εμείς πάντως συντάσσουμε ανακοίνωση, ήδη γίνονται τα εργαστήρια για να φτιαχτεί το σχέδιο του κώδικα ταξινόμησης που το σύστημα ακόμα στην αρχή θα είναι οικειοθελές. Εάν μπορέσετε να με βοηθήσετε να πείσω περισσότερους να υιοθετηθεί αυτό το οικειοθελές σύστημα, τότε θα κάνω και το επόμενο βήμα που θα είναι υποχρεωτικό. Θα ήθελα πολύ να δω αυτήν την όθηση στην πολιτική στην Ευρώπη που να προέρχεται από τις καταγγελίες των πολιτών, των καταναλωτών. Εάν δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να συμβάλλουν ευθέω στη διαμόρφωση της πολιτικής, δεν θα ε, προχωρήσουν. Στο, σχετικά με το switching, την αλλαγή δηλαδή και την ε, διαφάνεια, εγώ συμφωνώ με την ε, ιδέα αυτή η φραγμή στο switching είναι το ίδιο ζημιογόνιο όπως και η πραγματική φραγμή. Είναι λοιπόν και ένα θέμα διαπαιδαγώγησης. Θα αναφερθούμε και στις διάφορες α, πολιτικές που ακολουθούν ορισμένες βιομηχανίες ή σε ορισμένες αγορές με αθέμητο ανταγωνισμό και αλλού όπου πιέζονται οι καταναλωτές, pressure selling δηλαδή, για να αλλάξουν α, πάροχο. Συγχαίρω εν προκειμένου και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας επειδή προώθησαν την οδηγία, προώθησαν την οδηγία για να μπορέσουμε να βασιστούμε σε πλήρη εναρμόνιση και σε όλους τους τομείς πολιτικής να φτάσουμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο με χρήση όλων των μηχανισμών για την καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών ανταγωνισμού. Για την πρόταση του κυρίου Μάντερς. Ένα κουτί υποδείξεων δηλαδή. Θα το συζητήσω με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Καταναλωτών. Εγώ εννοώ, ε, λέει ο κ. Μάντερς χωρίς μικρόφωνο, τους ε, απλούς καταναλωτές. Ναι, αν όμως η, η ε, ε, το αναλάβει αυτό, απαντά η Επιτροπή και βέβαια ο καταναλωτής και η προστασία του μέσα στην οικονομική κρίση είναι μέρος της, της ατζέντα μας. Δεν μπορώ ωστόσο να σας δώσω υποσχέσεις που δεν θα τηρήσω μετά. Είναι και κάπως περιορισμένοι οι πόροι που διαθέτει η Γενική μου Διευθυνσή. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε θα μπορέσω να βρω πολύ προσωπικό για να εργαστεί πάνω στην ιδέα αυτή του κουτιού υποδείξεων. Πάντως είναι καλή ιδέα και είναι και καλή και για την προεκλογική εκστρατεία. Κύριε Νιούτον, ήταν Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Οι δύο ερωτήσεις μου είναι εξή. Είμαστε ακόμη μόλις στο δεύτερο έτος. Αλλά κατά πόσο θεωρείτε ότι το κοινό γνωρίζει τα, για τα θέματα που είπατε. Και δεύτερο, τα μέλη του Συμβουλίου συνεργάζονται μαζί σας ή, ανθίστανται μάλλον και λένε άλλη μια ε, ε, ιδέα που μας δυσκολεύει από τις Βρυξέλλες. Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ίσως τις πρωτεύουσές μας. Κύριε Αγγελάκα. Να ευχαριστήσω και εγώ την Επίτροπο για την παρουσία της και να τη συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Έχω μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί... Ah, you don't have translation. I can say it in English if you want. Okay. Again, I welcome you and I congratulate for the, the good job that you are doing. I have a very specific... Έχω λοιπόν μια συγκεκριμένη ερώτηση να σας υποβάλω. Είδαμε μετά, μετά από τον Σεπτέμβριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τις κυβερνήσεις των χωρών μελών. Είδαμε να παίρνουν μέτρα για να στηρίξουν το τραπεζικό σύστημα και τις τραπεζικές υπηρεσίες. Στο βαθμολόγιο σας έχετε δει να αυξάνεται ο ρυθμός των καταγγελιών των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις σχέσεις τους με το τραπεζικό σύστημα. Το ρωτώ αυτό διότι είδα σε διάφορες εφημερίδες διαφόρων χωρών μελών να αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πιέσουν, να σπρώξουν τα τραπεζικά συστήματα να συνεργαστούν, να δώσουν δάνεια να ε, συζητήσουν με πολίτες και εταιρείε επιχειρήσεις. Εσείς είδατε καμία αλλαγή, είδατε καμία αύξηση των καταγγελιών μετά από τον Σεπτέμβριο του 2008. Εσείς κύριε Λέχνερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο. Ήταν ενδιαφέρουσα η έρευνα με εντυπωσίασε θετικά το γεγονό ότι η κυρία Κούνεβα μίλησε κατά επανάληψη για τον ανταγωνισμό. Όπου δηλαδή δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμό, διαπιστώνει ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών, των καταναλωτών, είναι και μεγαλύτερη. Άρα τελικά ο ανταγωνισμό ωφελεί τον καταναλωτή. Όπω είπε όμω και η κυρία Βάιλερ προηγουμένω, στην ενέργεια είναι πολύ σημαντικό ο ανταγωνισμό. Στο τρένο και στο ε, λεωφορείο, ο ανταγωνισμό κάπου κάποια στιγμή θα καταλήξει σε κάποια σύνορα, σε κάποια, συγνώμη, σε κάποια όρια. Δεν θα μπορεί να προχωρήσει περισσότερο. Αλλά για τι τράπεζε θα πρέπει ε, να λειτουργεί ο ανταγωνισμό. Έχουμε και ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων. Με ενδιαφέρει, εάν βέβαια μπορείτε, δεν ξέρω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν και διάφορε ευαισθησίε ε, των διαφόρων χωρών, αλλά στι χώρε μέλη έχουμε διαφορετική πυκνότητα των ε, ε, τραπεζικών ιδρυμάτων, των πιστοτικών ιδρυμάτων κ.ο.κ. διαπιστώνεται διαφορές όπου δηλαδή υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών. Και όπως είπε και ο κύριος Αγγελάκας, η παρούσα οικονομική κρίση έχει περάσει στις, στις ερευνές έχει, έχει ληφθεί υπόψη και τι έχει προκύψει από αυτήν. Και Νομίζω οι αλλαγές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μελών έχουν καλώς. Υπάρχει έτσι και ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών. Δεν θα πρέπει να αντιστήξουμε. Ε, Γιατί ο κουτί υποδείξεων, αυτό δεν είναι κακή ιδέα. Υπάρχουν ήδη οι βουλευτές που παίζουν το ρόλο αυτό και εισπράττουν τα παράπονα ή τις καταγγελίες. Ας παρακολουθούμε λοιπόν τις καταγγελίες αυτές, ας ε, τις αναλύουμε, ας ε, πιέζουμε ώστε να επιληθούν τα προβλήματα, αλλά ας αφήσουμε τις καταγγελίες να τις χειρίζονται τα εθνικά επίπεδα. Και το ευρωπαϊκό επίπεδο ας κοιτάξει να προωθήσει τον ανταγωνισμό και μεταξύ των χωρών μελών. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα του κυρίου Νιούτον, είναι πολιτικής υφής. Ο πίνακας επιδόσεων δεν είναι νομοθετική πρωτοβουλία, δεν είναι δημοσκόπηση, είναι ένα πολιτικό μέσο και είναι σημαντικό για όλους μας να κατανοήσουμε ότι αν υπάρχει το σωστό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, που είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης, η αγορά θα δώσει ό,τι καλύτερο έχει για τον καταναλωτή. Βλέπουμε ότι δυστυχώς υπάρχουν, υπάρχει μια συμπεριφορά κατά του ανταγωνισμού και πρέπει να την εποπτεύσουμε γιατί οι καταναλωτές δημιουργούν το 58% του ΑΕΠ στην Ευρώπη που είναι πολύ μια πολύ μεγάλη εισρωή και γιατί θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβασης για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Διότι αν δεν υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβασης, τότε αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις ως προς την χρηματοοικονομική κρίση. Νομίζω ότι ο πίνακας επιδόσεων ε, αφορά εμάς τους ίδιους και δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς μεταχειριζόμαστε τον καθένα ως καταναλωτή. Και όπως είπε η κυρία Βάλ, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον στην αίθουσα τύπου όταν εξήγησα περί τίνος πρόκειται για τον πίνακα αυτό επιδόσεων. Γι' αυτό μεταφράστηκε και σε όλες τις γλώσσες και γι' αυτό συζητείτε εδώ και όταν μεταβαίνω στα κράτη-μέλη μιλώ με τις ενώσεις καταναλωτών και όχι με τους συναδέλφους. Καλό πράγμα η νομοθεσία, αλλά χρειάζεται και μία αίσια έκβαση. Και ε, πάντα προβάλλω τα διάσυστα στοιχεία που έχω έτσι ώστε οι άνθρωποι να γίνονται ε, να πιστεύουν περισσότερο, να έχουν μεγαλύτερη πίστη, διότι η πίστη είναι το καλύτερο νόμισμα της σύγχρονης οικονομίας. Είναι το καλύτερο αντίτιμο όταν μιλάμε για θέματα εσωτερικής αγοράς. Αν όμως δεν αποκτήσουμε αυτή την ε, ε, πίστη, δεν θα καταφέρουμε και πολλά στην αγορά. Δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Κανένας δεν θα αμελήσει τον ε, πίνακα αυτό και με την ε, δική σας βοήθη. Και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ένας ε, διεθνής φορέας για να μπορεί να έχει μια οπτική γωνία για όλες τις εθνικές κυβερνήσεις. Το θέμα αφορά και τον ανταγωνισμό και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Γι' αυτό μίλησα για χώρες με καλές επιδόσεις και ε, χώρες με χειρότερες επιδόσεις. Δεν θέλουμε να κατονομάσουμε κανέναν. Θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη εσωτερική αγορά με καλύτερο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης. Άρα ο ανταγωνισμός είναι στα γονίδια μας. Γι' αυτό θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για αύξηση ανταγωνισμού στο Συμβούλιο. Θα υποβάλω το θέμα στους Υπουργούς και ό,τι και να κάνω εγώ και οι συνάδελφοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τους υποστηρίξουμε αυτή την ανάλυση της αγοράς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Αγγελάκα και λέει ευχαριστώ πολύ η Επίτροπο στα ελληνικά. Στη σελίδα 22 και 9 εδώ έχουμε ειδικά στοιχεία για τον τραπεζικό τομέα. Έχουμε 50 αριθμητικά στοιχεία και συγκρίσεις και εδώ έχετε το στοιχείο 20 όπου τα τραπεζικά τέλη ε, αναγράφονται αναχώρα ανάλογα με το προφίλ που επιλέγουμε. Έχουμε την Ελλάδα λοιπόν εδώ η οποία δυστυχώς είναι έχει τις χειρότερες επιδόσεις. Με συγχωρείτε που πρέπει να σας το πω, αλλά μπορείτε να συγκρίνετε τουλάχιστον και να πιέσετε κάπως γιατί είναι ένα μέσο στα δικά σας χέρια και στα δικά μας χέρια. Η Ελλάδα θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα και το ελπίζω, το εύχομαι ολόψυχα. Άρα πρέπει να επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος για την αύξηση της διαφάνειας στα τραπεζικά τέλη και στην παροχή συμβουλών. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Και υπάρχει η χρηματοπιστωτική κρίση Άρα μιλάμε για μετά τον Οκτώβριο, δεν ξέρω κατά πόσο τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα μετά τον Οκτώβριο. Αλλά ήδη τον Οκτώβριο ήταν πολύ αργά, γιατί κλείναμε τα στοιχεία και τα αναλύαμε. Κύριε Λάκνερ, έχουμε ε, λεπτομέρειες αναχώρα, ανάλογα με τις αγορές. Θέλουμε να συγκρίνουμε τις χώρες Οι χώρες θα πρέπει να ανταγωνίζονται στην αγορά για την αγορά που είναι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις παράλληλα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να πείσω τις χώρες ότι θα πρέπει να μας δώσουν στοιχεία. Έπρεπε να δώσω μάχη, αλλά τελικά τα κατάφερα και είμαι ευγνώμων προς τον Επίτροπο Αλμούνια, ο οποίος ήρθε σε επαφή με την Eurostat για συνεργασία και είναι μια κοινή προσπάθεια αυτή της Επιτροπής. Πολύ και πολύ καλή ομαδική εργασία. Η κυρία Ρόιτοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Επίτροπε, κυρία Επίτροπε που ήσασταν μαζί μας. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι ευρέως ορατή η εργασία σας και ευεργετή τους Ευρωπαίους πολίτες και καταναλωτές. Χαίρομαι που ορίσατε την ενέργεια ως πρωτοβουλία ε, λίγους μήνες πριν. Και ξέρετε ότι λίγους μήνες πριν επίσης μιλήσαμε για το τρίτο πρόγραμμα ενέργειας Ξέρετε ότι ελήφθησαν υπόψη προτάσεις ε, αυτής της Επιτροπής για την Προστασία των Καταναλωτών. Ορισμένα μέτρα είπατε ότι θα είναι δική σας προτεραιότητα, όπως η αλλαγή παρόχου. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, μετά την ε, διενέργεια έρευνας, ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια του χαμηλού ρυθμού αλλαγής ε, παρόχου. Επίσης ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει και η εναρμόνιση των τιμολογίων. Η ενιαία θηρίδα δικαιοδοσίας για τις καταγγελίες καθώς και οι χαμηλότερες τιμές για ορισμένους, ε, για καταναλωτές, δηλαδή ευπαθείς ε, κατηγορίες. Ο ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο για τα δύο νέα κράτη-μέλη, Βουλγαρία και Ρουμανία, υπάρχουν ε, στατιστικά στοιχεία. Και μια άλλη ερώτηση εκεί όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει μία ε, εταιρεία, ένας πάροχος ε, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πώς μπορούμε να παρέμβουμε, πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, διότι από όσο ε, γνωρίζω τα πρόστιμα είναι πολύ χαμηλά. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσετε για να τηρηθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και σε περίπτωση ολιγοπολίων θα πρέπει να ε, δούμε ε, πώς μπορούν να ευεργετηθούν οι καταναλωτές που μπορεί να είναι μια πολύ υψηλή κατηγορία. Ως προς τις καταγγελίες ξέρουμε ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα. Αυτό αφορά και τις μη κυβερνητικές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ε, ατζέντα Πολλές φορές ε, δεν υπάρχει παρά μία τηλεφωνική γραμμή, δεν υπάρχει hotline, δεν υπάρχει μία 24ωρη υπηρεσία, υπηρεσία και δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πώς ε, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε ε, αυτές τις μη κυβερνητικέ έτσι ώστε να έχουν μόνιμη τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστώ. Merci, Madame la Ευχαριστώ που ήρθατε να ανταλλάξετε απόψεις μαζί μας, διότι είναι ένα θέμα ύψης της ε, σημασίας να εστιάσουμε την προσοχή μας στις ίδιες μας τις χώρες για να τα καταφέρουμε καλύτερα. Έχω ένα ερώτημα για να συμπληρώσω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι. Δηλαδή, αναμένοντας ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης, ε, πολλές χώρες ε, είδαμε ότι δεν ε, τηρούν την εποπτεία της αγοράς για να, δούμε, για να δουν πού δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός για να βοηθήσουν τους καταναλωτές, αλλά λήψη ενός ενιαίου ε, συστήματος ταξινόμησης, παρόλο που κατονομάζουμε ε, ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων ε, και η Γαλλία ως προς την κινητή τηλεφωνία και την έλλειψη ανταγωνισμού σε ορισμένες περιοχές και διοικητικά διαμερίσματα Ήδη σήμερα, ακόμα και σήμερα, στην εκλογική περιφέρεια υπάρχει μια μεγάλη ε, κοινωνική αναταραχή γιατί το θέμα δεν εντοπίστηκε εγκαίρως. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί η Γαλλία έχει κατηγορηθεί σε πολλούς τομείς. Πώς μπορούμε όμως να ασκήσουμε πίεση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα έμπρακτα τη στιγμή που δεν ε, έχουμε επιφέρει λύσεις. Αναφέρω, αναφέρομαι σε τρεις τομείς. Η έλλειψη ανταγωνισμού στην ε, κινητή τηλεφωνία δεν αφορά μόνο τα τηλέφωνα, όπως είπε και ο συνάδελφος, αφορά το, τα ευρυζωνικά δίκτυα, αλλά και την, και την τηλεόραση, τα, την πρόσβαση στα δίκτυα γενικότερα. Γιατί τα ευρεία δίκτυα διανομής δεν ανταποκρίνονται σε επίπεδα που θα επιθυμούσαμε. Και πολλές φορές έχουμε μονοπόλια και ολιγοπόλια, άρα δεν μπορεί να υπάρξει απελευθέρωση τιμών. Ένας άλλος τομέας που είναι πολύ σημαντικός είναι το κόστος μεταφοράς για να φτάσουμε σε μία σταθεροποίηση και να μειωθούν οι τιμές με τα δίκτυα ευρείας διανομής. Πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε κρατικό επίπεδο έτσι ώστε να ασκήσουμε έμπρακτα πίεση, διότι όλα τα μέσα θεωρητικά είναι πολύ καλά, αλλά δεν έχουν κανένα μεγάλο αντίκτυπο στο τι θα έπρεπε να κάνουμε στο μέλλον. Άρα είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, κατάσταση η οποία ισχύει στην πράξη. Κυρία ε, Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να ρίξω μία μικρή βόμβα ή χειροβομβίδα, αν θέλετε, στη συζήτηση, διότι ο, ο πίνακας είναι πολύ καλός για να αντιμετωπίσουμε ε, ειδικά ζητήματα. Αν δούμε τον τομέα της αγοράς ενεργείας, Βλέπω ότι αναμείναμε πολύ χρόνο για δράση σε αυτό το τομέα και είχαμε μία δυνατότητα με την πρωτοβουλία του τρίτου πακέτου ενέργειας και η εισηγήτριά μας έκανε πολύ καλή εργασία κυρία Νέρης και νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε μία ε, χάρτα καταναλωτών ή ένα checklist. Ο κύριος Πίμπαλξ δεν ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο γιατί δεν θα είχε νομική ισχύ. Αλλά υπάρχουν πολλοί τομείς όπου θα μπορούσε να προωθηθεί μια νομοθετική δράση. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Αναμείναμε επί μακρόν και νομίζω λοιπόν ότι ο καταναλωτής χάνει την εμπιστοσύνη του στην Ευρώπη. Εγώ βρέθηκα σε μια διάσκεψη με ε, οργανώσεις καταναλωτών όπου συζητήσαμε το πακέτο ενέργειας στο Λονδίνο όπου μια ένωση καταναλωτών μίλησε για καλύτερη πληροφόρηση και περισσότερα δικαιώματα. Και αυτά τα σημεία εσείς ε, θίξατε και στον πίνακα, δηλαδή ε, διαφάνεια, συστήματα ADR έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να διαμαρτυρηθεί και να καταγγείλει αυτό το τιμολόγιο. Και εγώ πρόβαλα ένα σχέδιο δράσης 10 σημείων. Ο κύριος Πίλπαξ μου είπε ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει νομοθετικού περιεχομένου ε, προτάσεις όπως το, τη λίστα ελέγχου. Ως προς τον ανταγωνισμό και την ε, ανοιχτή αγορά, εδώ αντιτάχθηκε σε μια νομοθετική πράξη. Βεβαίως υπάρχουν ανοιχτές αγορές και απελευθέρωση, αλλά αν υπάρχει ε, μια καταγγελία από μια μικρή οργάνωση που χρησιμοποιεί ε, μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ως μικρή οργάνωση και έχει έναν πάροχο από τη Γερμανία και ζητά ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο με διαφάνεια, μετά ε, από πέντε χρόνια ε, λάβανε ένα τιμολόγιο για 7.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να επιληθεί αν υπάρχουν τιμολόγια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Άρα ε, θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και ο Επίτροπος Ρυθμάτων Ενεργείας είναι αρμόδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να αποφανθείτε και να φτάσετε σε απτά αποτελέσματα. Πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτές τις προσδοκίες, διότι έχουμε υψηλές ε, προσδοκίες από τον πίνακα επιδόσεων. Έχουμε λάβει πολλές καταγγελίες από το εκλογικό μας ε, σώμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε μέσα διεκπαιρέωσης και πολλές φορές οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν δράση και αναρωτιέμαι τι μπορείτε να κάνετε γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έναν πίνακα επιδόσεων, έχουμε αναγνωρίσει τα προβλήματα, έχουμε υποβάλει τροπολογίες, αλλά δεν έχουμε ε, απτά αποτελέσματα. Δείτε το και στην κινητή τηλεφωνία. Ακολουθήσαμε την ομοθετική οδό στο τέλος, αν και πολλοί θεώρησαν ότι ο βιομηχανικός τομέας και η αγορά θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν από μόνοι τους, αλλά δεν έγινε και πολλές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αντιτάσσονται στη νομοθεσία, δηλαδή δεν υπάρχει υποστήριξη από την βιομηχανία. Και αυτό αφορά και τα SMS ή την πρόσβαση στο διαδίκτυο τηλεφωνικός. πώς μπορούμε να έχουμε άμεση ε, δράση. Γιατί αν η βιομηχανία mm. δεν συμφωνεί, δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι καταναλωτές. Και ο Μάλκομ έχει μία ερώτηση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την Επίτροπο γιατί δεν ήμουν εδώ εξ αρχής, αλλά σας είπα ότι έπρεπε να βρεθώ στον ε, τριμερή διάλογο για τις τηλεπικοινωνίες, για το πακέτο και αυτό σε σχετίζεται με αυτό που προελέχθη δηλαδή ο σύνδεσμος με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές διότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν άμεση ευθύνη και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουμε μία χάρτα ε, υπέρ του καταναλωτή που έγινε δεκτή στο πακέτο που υπάρχουν ε, κοινά, κοινά πρότυπα σε σχέση με την αλλαγή παρόχου και την τιμολόγηση. Ε, μιλήσατε και για την κάλυψη, τα δίκτυα κάλυψης ως προς την ε, κινητή τηλεφωνία, αλλά πώς ε, το αντιμετωπίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες και να αποφασίζουν ποιες αλλαγές πρέπει να επέλθουν. Η αγορά της ενέργειας δεν είναι ομοιογενής, αλλά ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό έδαφος για να δούμε πώς ανταποκρινόμαστε στα ζητήματα που εφήγησαν. Αυτά είναι τα τελευταία ερωτήματα προς την Επίτροπο. Ίσως θέλετε να ανακεφαλαιώσετε η Επίτροπος. Θα ξεκινήσω με την κυρία Γέτουβα θα απαντήσω στα αγγλικά αν μου το επιτρέπετε. Αλλά φυσικά μπορούμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας αργότερα στην Βουλγαρική. Οι βασικοί λόγοι για την μη αλλαγή παρόχου αναφέρομαι για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, αλλά στην Βουλγαρία είναι το κόστος της αλλαγής διότι οι καναλτές δεν κατανοούν πολλές φορές τις προσφορές και δεν μπορούν να κάνουν την απαραίτητη σύγκριση και διότι θεωρείται, εκλαμβάνεται μάλλον ως κάτι περίπλοκο και δύσκολο. Τώρα στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβάνουν και της Βουλγαρίας, δεν υπάρχουν εκστρατείες ενημέρωσης, πολλές φορές δεν διαβάζουμε καν τους, τα τιμολόγια και φυσικά δεν κάνουμε σύγκριση ανάμεσα τα τιμολόγια. Ως εκ τούτου πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας και το πρώτο βήμα κατά την άποψή μου είναι να καταστεί η τιμολόγηση πιο εύπεπτη. Διότι έτσι οι άνθρωποι θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, αφού φυσικά κατανοήσουν τι περιέχουν τα τιμολόγια. Εγώ βρίσκομαι πάντα σε αγώνα εναντίον στους παρόχους και την επόμενη εβδομάδα θα τους ξανασυναντήσω. Έχω υπογράψει ένα είδος μνημονίου συνεννόησης προκειμένου να καταστήσουμε, να προωθήσουμε μια εκστρατεία ενημέρωση. Δυστυχώ, οι προσπάθειες μέχρι τώρα δεν έχουν στεφθεί υπό επιτυχία, αλλά στο επόμενη εβδομάδα προσπαθήσω να το πετύχουμε. Αυτό που προτείνεται για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το καράπο θα μπορούσε να βοηθήσει στο να βελτιώσει το επίπεδο κατανόηση σε θέματα προστασία καταναλωτή ανά την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένη και τη Βουλγαρία φυσικά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοηθούμε για να δούμε προχωρήσουμε. Τώρα για τις ε, καταγγελίες των καναλωτών μπορούν να εναρμονιστούν σε ε, κοιοθελή βάση και θα ήθελα η Βουλγαρία να συμμετάσχει σε αυτό το έντυπο της, ε, για τις καταγγελίες της Λούτερ. Δεν υπάρχει έρευνα αναχώρα. Εδώ Μιλάμε για αγορές και όχι για χώρες. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε ένα κεφάλαιο για τη Ρουμανία, αλλά θα έχετε ένα κεφάλαιο για τις ε, ε τραπεζικές προμήθειες ε, κλπ. Και θα δείτε λοιπόν πού βρίσκεται η Βουλγαρία. Τώρα για τα hotlines ε, κλπ. που θίξατε. Εάν έχουμε έναν πάροχο, όπως είπατε, στην ηλεκτρική ενέργεια ή οπουδήποτε αλλού. Και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να είναι τριπλά πιο προσεκτική. Χρειαζόμαστε να υπάρχουν οργανώσεις καταναλωτών που θα συνεργάζονται και να παρατηρούν πώς υπολογίζονται οι τιμές, πώς γίνεται η τιμολόγηση και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπάρχει υποχρέωση για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ και από σας και από τις εθνικές αρχές να εξετάσετε το ζήτημα και να δείτε τι ρόλο παίζουν οι καταναλωτές σε αυτήν την ρύθμιση των τιμών στις περιπτώσεις όπου το υπάρχει μονοπόλιο. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για τα μονοπόλια ε, στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και την βελτίωση του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός είναι ένας ε, πυλώνας της εσωτερικής αγοράς και μία από τις βασικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ πως αυτά που έχουμε εδώ είναι έλλειψη επιβολής ε, του νόμου, έλλειψη συμμόρφωσης. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο από το να δηλώσω εκ νέου ότι η συμμόρφωση είναι θέμα κράτους μέλους. Δεν έχουμε μία ε, αστυνομία καταναλωτή, δεν μπορούμε να, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε να στείλουμε κάποιους για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους σε κάθε κράτος μέλος. Εντάξει, αν υπάρχουν κάποια επικίνδυνα τρόφιμα, επικίνδυνα αγαθά, εντάξει, τώρα μπορούμε να Αλλά για την επιβολή των ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών, αυτό απόκειτο σε κράτη-μέλη. Το που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να ε, ε, αλληλοενημερωνόμεθα για το πώς έχουν τα πράγματα, ποιες είναι οι εξελίξεις. Πέρυσι διοργανώσαμε το πρώτο ε, φόρουμ πολιτών για θέματα ενέργειας, αλλά αυτό ήταν ένα φόρουμ. Ενημερώνουμε, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς αυτή την υποχρέωση για, σε ό,τι φορά τους ε, πίνακες επιδόσεων, αυτό είναι κάτι το οποίο μας δείχνει την, ε, κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες, ε, τι αποτέλεσματα δίδουν οι καταγγελίε τους κλπ. Στο μέλλον θα μπορούσα να σκεφτώ, εάν δεν υπάρχει, δεν ασκούνται αυτά τα δικαιώματα, τότε να υπάρχει προσφυγή επί παραβάσεων και να επιβάλλεται κάποια κύρωση, ένα πρόστιμο, επειδή το κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται, δεν επιβάλλει τον, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία προκατασκευασμένη απάντηση. Εγώ θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου, αλλά δεν μπορώ να σε επισκεφθώ ότι θα υποκαταστήσω τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες. Εάν θα μπορούσα να το πράξω, πιστέψτε με ότι θα ξεκινά <clears throat> με τη χώρα την οποία γνωρίζω καλύτερα. Και κυρία Γιώτοβα θα υπέβαλα τις απόψεις μου στις εθνικές αρχές της Βουλγαρίας. Τώρα, η ερώτησή σας σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε. Εάν συμφωνείτε με μένα, θα σας πρότεινα να διοργανώσουμε το φθινόπωρο ένα, μια ακρόαση. Θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε τις ρυθμιστικές αρχές. Ε, φυσικά, φυσικά, φυσικά εγώ είμαι πρόθυμη να συμμετάσχω. Επίσης, πρέπει να επανεφεύρουμε την επιβολή αυτών των κανόνων και τον τρόπο επιβολής στην Ευρώπη. Τώρα, η ρύθμιση των τιμών, αυτό που πράξαμε με το Ρώμα, την ε, περιαγωγή, είναι κάτι το σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να παροτρύνουμε την αγορά προτού να ακολουθήσουμε οποιαδήποτε άλλη λύση. Δεν ναι, θα αφιστούμε λοιπόν κόπον. Προτείνω τη διοργάνωση μιας ακρόασης και την ε, επιτήρηση βολής του, των νομοθεσίας. Συμφωνώ μαζί σας. Κάτι ακόμα από τον κύριο Χάρμπορ. Ικανοποίηση και ικανοποιητικό ποσοστό αλλαγής παρόχου. Υπάρχουν παράπονα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται ε, τα, οι εταιρείε αυτήν την, ε, τα αιτήματα η ικανοποίηση είναι χαμηλή για τα ε, τη σταθερή τηλεφωνία και οι προσφορές από τις εταιρείε τηλεπικοινωνιών είναι πιο εύκολα να αξιολογηθούν. Και στα δύο, στα δύο αυτά σημεία λοιπόν το επίπεδο του ο είναι καλός. Ε, ε, χρησιμοποίησαμε την οδηγία που ζητούσε κάποιες περαιτέρω προφορίες, αλλά βέβαια είμαι ικανοποιημένος για το switching. Εγώ θα συνεχίσω το διαπραγματεύσει έτσι ώστε η ταχύτητα αυτής της αλλαγής παρόχου να είναι μεγαλύτερη. Θα μπορούσε λοιπόν ε, αυτή η θερική εμπειρία που έχουμε στο τομέα των να τη μεταφέρουμε και στο τομέα τη ενέργεια. Το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η τιμολόγηση. Εντάξει, οι εταιρείε ε, μπορούν να λένε και να δηλώνουν ότι θα σας ε, υποβάλουν ένα αναλυτικό τιμολόγιο κάτι όμως που συνήθως δεν κάνουν. Όπως σας είπα, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εστιάσατε στους κλάδους που μας απασχολούν ιδιαίτερα, αλλά εμείς δεν θα πάψουμε να σας ε, στηρίζουμε και να σας προτείνουμε ιδέες για την βελτίωση της κατάστασης και φυσικά μπορούμε να σας υποστηρίξουμε και στο Σώμα των Επιτρόπων διότι δεν με εντυπωσίασε η προσέγγιση του κυρίου Φιλμπαξ στο θέμα της ενέργειας. Αυτή είναι η δουλειά του, είναι επίτροπος αρμόδιος για την ενέργεια. Αλλά δεν νομίζω ότι το πακέτο πρότεινε ικανοποιεί τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπουμε στο να σας ξαναδούμε σύντομα. Okay, Η Ας επανέλθουμε στα θέματά μας, στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως μας, ο συγγετής μας είναι παρόν. Θα συζητήσουμε για τον κανονισμό για τα ε, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον εισηγητή και μετά ε, στα μέλη που ενδεχομένως θα θέλουν να ομιλήσουν. Ο κύριος Καμάλ. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να, δούμε όλες, να δω όλες τις τροπολογίες, όπως άλλωστε πολλά μέλη μας εδώ, διότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση με τις μεταφράσεις. Πάντως ε, κάπως ε, τις κοιτάξαμε δεν με ευνηδίασαν οι τροπολογίες γιατί απηχούν ε, τις συζητήσεις που έγιναν και στην Επιτροπή μας αλλά και σε όλο το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό εξετάζοντας την πρόταση της Κομισιόν μπορεί να σκεφτεί κανείς είτε ότι είναι περιττή νομοθετική εργασία ή ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρή η Ευρωπαϊκή Επιτροφή ότι το κέρδος είναι κακό και ότι δεν πρέπει οι παροχοί τηλεφωνικών υπηρεσιών να αποκομίζουν κέρδος από τις υπηρεσίες που προσφέρουν και άρα πρέπει να τους φερθούμε πιο αυστηρά. Τώρα, εξετάζοντας το πώς θα προχωρήσω, προσπάθησα να συνεργαστώ με την Επιτροπή Βιομηχανίας τον εισηγητή της και τους σκιώδης εισηγητές οι οποίοι επιθυμούν να ακούσουν εμάς πρώτα για θέματα διαφάνειας, αφού εμείς είμαστε αυτοί που ηγούμεθα της εκστρατείας για την προστασία των καταναλωτών. Και προσπάθησα να ρίξω ιδιαίτερο φως με τις δικές μου στην προστασία του καταναλωτού και στην διαφάνεια. Και η Επιτροπή Βιομηχανίας, Ήτρε, θα ήθελε περισσότερο να ρίξει βάρος σε θέματα χονδρικής αλλά και λιανικής Σωστό είναι αυτό βέβαια και για τις δύο αυτές οι επιτροπές να τροπολογήσουν δηλαδή τα μέλη τους ό,τι επιθυμούν. Εγώ πάντως προσπάθησα να ρίξω ιδιαίτερα το βάρος στην διαφάνεια. Νομίζω ότι θα φανεί και από τις τροπολογίες μου ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι πελάτες αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκείς και νομίζω ότι είναι σημαντικό οι καταναλωτές να διαθέτουν την μέγιστη δυνατή πληροφόρηση όταν κάνουν περιαγωγή, ώστε να μπορούν να επιλέγουν εν γνώση ε, το, του τι θα ε, αναγκαστούν τελικώς να πληρώσουν. Είπα ότι δεν είναι αρκετό οι πάροχοι να λένε ότι κοιτάξτε αν θέλετε τις τιμές μας στο διαδίκτυο ή θα τις δείτε στην σύμβαση που υπογράψατε μαζί μας όταν ε, αποκτήσατε την σύνδεση. Δεν είναι σωστό αυτό. Το αντεπιχείρημα βέβαια είναι ότι οι πελάτες λαμβάνουν, δέχονται υπερβολικά πολλές πληροφορίες και αυτό το λένε και αυτοί που είναι υπέρ της ε, νομοθεσίας αυτής. Αλλά δεν θέλουμε να μπορούν να πούν οι καταναλωτές ότι δεν είχαν επαρκή πληροφόρηση. Ακόμα και αν είναι υπερβολική, είναι καλύτερο να είναι υπερβολική η πληροφόρηση παρά μην είναι επαρκής. Και ας επιλέξουν τέλος πάντων οι καταναλωτές τι επιθυμούν να κάνουν. Δεν νομίζω να χρειάζεται να πω σε άλλε λεπτομέρειε, γιατί οι τροπολογίε απηχούν πραγματικά τη συζήτηση όπως διεξήχθη εδώ στην Επιτροπή. Όπως συζητήσαμε λοιπόν μέχρι εδώ. Θα αρκεστώ σε αυτά για την ώρα και θα συνοψίσω πάλι στο τέλος τη συζήτηση, Η Πρόεδρος. Καλά κάνει ο εισηγητής και ρίχνει βάρος ε, στα θέματα που δεν είχαμε συζητήσει προηγουμένως που θα με συζητήσει ορισμένα θέματα όπως ε, τιμές ελιανικής για, του, πελάτη δηλαδή ή, και την κακή συνήθεια των παρόχων να αποκομίζουν κέρδος από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ας δούμε τώρα τι έχουν να πούν οι σκιώδεις συγκητές, ο κύριος Μπιφόν πρώτα που είναι των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο εισηγητής ξεκαθάρισε που βρίσκονται τα μέτωπα, ας πούμε έτσι. Εγώ συμφωνώ μαζί του ότι επί του παρόντος και λόγω του ότι λείπουν ορισμένες μεταφράσεις τροπολογιών δεν μπορούμε να τις συζητήσουμε όλες σε βάθος. Εγώ συγκαταλέγομαι περισσότερο μεταξύ εκείνων, στον τομέα αυτό δηλαδή, όπου θεωρούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή βάση για συζήτηση. Κάτι που δεν είναι αρκετά αυστηρό ωστόσο για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που ε, καταθέσαμε, ο στόχος μας ήταν να αυξήσουμε κατά το δυνατόν την προστασία των κατανολωτών. Υπάρχει ένα πλήθος δυνατοτήτων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ωστόσο σε μια κοινή προσπάθεια και με τον εισηγητή. Η κυρία Γιώργινσεν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω ε, δανέζικα. Δεν είμαι κομμουνίστρια, ελπίζω να φερθώ και να ηχήσω ως φιλελεύθερη. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε ήδη συζητήσει ορισμένα από τα θέματα αυτά στο παρελθόν. Θέλω να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα άπαξ και διαπαντός. Στον τομέα αυτό είμαι φιλελεύθερη. Δεν επιζητώ ρυθμίσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις ως αυτοσκοπούς. Έχω καταθέσει ορισμένες τροπολογίες. Με τον κύριο Καμάλ συζητήσαμε δύο θέματα. Το λεγόμενο value pricing και το water bed effect. Δηλαδή τον κίνδυνο με την περιαγωγή να ανεβοκατεβαίνουν τιμές, δηλαδή να μειωθεί στην περιεγωγή, να αυξηθούν όμως σε άλλα, όπως εθνικά SMS και τα λοιπά προϊόντα. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, διότι, διότι και εκεί ισχύει ο ανταγωνισμός. Πρόκειται για αγορά η οποία λειτουργεί στη βάση των συνήθων αρχών της αγοράς εφόσον ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει, θα επιλέξει για τον ΑΒ λόγο μία εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών στην βάση του τιμολογίου της. Ω συνέπεια του ανοίγματο της αγοράς περιαγωγής μπορεί ενδεχομένως να οδηγηθούμε στο άνοιγμα των εθνικών αγορών ώστε να εξηγιανθούν όλες οι αγορές αυτές. Και αυτό είναι βεβαίως το, ε, η βάση της φιλελεύθερης πολιτικής που με ενδιαφέρει γιατί είναι υπέρ του, ε, των συμφερόντων των καταναλωτών όπως είναι και υπέρ των συμφερόντων του κλάδου. Και σε ό,τι αφορά το λεγόμενο value pricing, εγώ θεωρώ ότι οι αγορές θα λειτουργήσουν μόνο εφόσον η προσφορά είναι ελεύθερη και εφόσον ο καταναλωτής έχει την ελευθερία να επιλέξει. Σχετικά τώρα με τις τροπολογίες μου. Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας και κυρίως να επιτευθούν τα ποθούμενα αποτελέσματα. Οι συνάδελφοί μου εδώ στην Επιτροπή μας μίλησαν και για την περίφημη sunset clause εν προκειμένου. Εγώ δεν είμαι απόλυτα πεισμένη ότι έχουμε εν τέλει επιλέξει την σωστή διατύπωση για αυτή την sunset clause και γι' αυτό εγώ ίδια δεν έχω προτείνει τίποτα σχετικό. Εάν ωστόσο κατατεθεί πρόταση που θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική, τότε είμαι διατεθειμένη να την συζητήσω. Και επίσης αυτά τα price caps, αυτές οι ε, ανώτατες τιμές της Επιτροπής, βρίσκω ότι εξακολουθούν και είναι πολύ υψηλές και δεν είναι σε καμία σωστή αναλογία με τις δαπάνες. Τώρα, το άλλο θέμα, ε, το λεγόμενο bill shock, ξαφνικά δηλαδή ο καταναλωτής λαμβάνει ένα τεράστιο λογαριασμό και ε, δεν γνωρίζει από πού βγαίνουν όλα αυτά τα έξοδα, όλες αυτές οι, ε, όλα αυτά τα υψηλά τέλη. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να έχουν μια πλήρη εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα cut-off limit εγώ όμως δεν το βρίσκω αυτό ικανοποιητικό. Θα πρέπει να δοθεί, αφόσον ε, δοθεί η δυνατότητα αυτή στους καταναλωτές να ε, έχουν μια σύνδεση με ένα cut-off limit, θα πρέπει να το γνωρίζει ο καταναλωτής και να έχει και την γνώση, να είναι δηλαδή προφορημένος και πώς μπορεί να υπερβεί αυτό το cut-off limit, αυτό το ανώτατο όριο. Στην πολιτική μου πάντως ομάδα Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές γνώμες. Θα έλεγα μάλιστα ότι κινδυνεύουμε να έχουμε και περισσότερες γνώμες από, ό,τι, από όσα είμαστε μέλη. Ε, αυτό ίσως είναι χαρακτηριστικό των φιλελεύθερων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εδώ, καθώς θα πλησιάζουμε και στην ψηφοφορία. Θα αναζητήσουμε και στη δική μου πολιτική ομάδα κάποιο τρόπο βέβαια να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Αντίθετα με τους φιλελευθέρους εμείς δεν καταθέσαμε τροπολογίες διότι μας ικανοποιεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προσθήκες, οι συγκλώσεις του κυρίου Καμάλ σε σχέση με μια προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης διαφάνειας μας βρίσκουν σύμφωνους και θα τις υποστηρίξουμε. Στη Γερμανία αντιμετωπίζουμε ακόμη προβλήματα με ορισμένους providers. Πάντως οι τροπολογίες κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε και έχουμε και δυνατότητα να επιλέξουμε μεταξύ των τροπολογιών αυτών. E, έχω ορισμένα θέματα σχετικά με την περιαγωγή που με απασχολούν. Νομίζω ότι ο εισηγητής ε, γνωρίζει τις ε, προτάσεις μου. Δεν συμφωνώ με την στάση εκείνη που λέει ότι η πρόταση της Επιτροπής για τα price caps πρέπει να απορριφθεί. Οι καταναλωτές υποτίθεται ότι πρέπει να διαθέτουν, να έχουν διαφάνεια δηλαδή και ε, προστασία για την περιαγωγή. Εγώ θέλω να υπάρξει περισσότερος ανταγωνισμός όπου, που να οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Εγώ θα προτείνω λοιπόν να ε, επιβληθούν price caps και εκτός από αυτό Νομίζω ότι οι προτίσει που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τιμέ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξακολουθούν να είναι υψηλέ. Υπάρχει ακόμη περιθώριο για μείωση των τιμών, για παράδειγμα για τα γραπτά μηνύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει 11 λεπτά. Εγώ θα προτείνω 9 λεπτά. Νομίζω ότι είναι σωστή η ιδανική τιμή. και από 4 σε 2 για τις χοντρικές τιμές όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Τροπή. δηλαδή 4, εγώ θα προτείνω 2 μεταξύ των ε, ε, εταιριών επομένως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει και ορισμένα μέτρα για την ε, διασφάλιση τη διαφάνεια, της διαφάνειας των τιμολογίων που λαμβάνουν οι καταναλωτές, το οποίο ωφελεί βέβαια τους καταναλωτές, έχω ορισμένους ε, ορισμένες αμφιβολίες ε, σχετικά με, τις, ε, την επιρροή των τιμών χονδρικής επί των τιμών λιανικής σχετικά με την μετάδοση δεδομένων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Όλε Σμιτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μαλώσω με την αγαπητή μου συνάδελφο κυρία Ρίς Γιώργενσεν. Συνήθως δεν διαφωνούμε Έχω όμως ορισμένες θεμελιώδεις ερωτήσεις, κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θεωρώ, όπως είπε και ο εισηγητής, ότι μπορεί όντω να είναι ένας ολιστηρός κατήφορος. Θα ήθελα ε, να ακούσω λιγάκι τι έχει συζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην περίπτωση αυτή και ποια ίσως, τα, ποια ίσως θα είναι τα επόμενα θέματα σχετικά με τις υψηλές τιμές διότι ο βασικός λόγος που αντιδράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για να προστατεύσει τους καταναλωτές. Εγώ νόμιζα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακα των συνθήκων προσπαθεί να προστατεύσει και την ελεύθερη αγορά που αποτελεί θεμέλιον μάλιστα και των κριτηρίων της Κοπενχάγης αγαπητή κυρία Ρίση Γιώργενσεν. Δεν προσπαθώ βεβαίως να θίξω κανέναν εδώ αλλά ε, εντυπωσιάζομαι που ακούω ορισμένα πράγματα, διότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι κάποια άλλα προϊόντα που να έρθετε και να μας πείτε ότι είναι υπερβολικά ακριβά και ε, ίσως έχουν ε, και άλλες κακές πτυχές. Τουλάχιστον γιατί εμείς οι πολιτικοί βέβαια μπορούμε να αντιδράσουμε πιο απότομα και ίσως και να πούμε τη μια εβδομάδα ένα πράγμα και την επόμενη εβδομάδα κάτι άλλο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι και η ευθύνη της να δρά στη βάση αρχών. Δεν μπορεί να πει απλώς ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, το λύνουμε με μια οδηγία και λέμε στους καταναλωτές όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Κοιτάξτε κύριοι σας, προστατεύουμε. Να, πέφτουν οι τιμές. Γιατί εγώ θεωρώ ότι το επιχείρημα είναι λάθος, μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω σε ποια σε ποιε αρχές, σε ποια κριτήρια βασίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι είπατε? ενδιαφέρον αυτό το επιχείρημα των αριστερών ή των πρασίνων, λέει ο κ. Σμιτ. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, θα πω ότι ως φιλελεύθερος μπορείτε να σκέφτεστε ταυτόχρονα πολλά πράγματα με το, με το, ένα μυαλό που έχετε. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς. Δεν άκουσα τι είπε η συνάδελφός μας εκρηξιών σας. Αλλά ο μόνος τρόπος για να δικαιολογήσουμε την ύπαρξή μας είναι να βασιστούμε στην ε, συνθήκη και η συνθήκη προβλέπει και προστασία των καταναλωτών και ελεύθερη αγορά. Είμαι βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει τις δικές της ιδέες, αλλά πρώτα θα ακούσω τον κύριο Χάρμπορ for this approach, Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε δύο σημαντικά μέτρα που αναγράφονται εδώ και που αντικατοπτρίζουν τις συμφωνίες μας εδώ στην Επιτροπή σε σχέση με τα δικαιώματα των Χριστών. Και νομίζω ότι θα πρέπει να σας επισύρω την προσοχή σε αυτό. Καταρχήν θέλουμε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τους ε, καταναλωτές, να τη διασφαλίσουμε αυτή. αν ε, ο πάροχος ε, περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και εδώ μιλάμε για υπηρεσίες τύπου Skype ή φωνητικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο και αυτό θα πρέπει να το ξέρουν οι καταναλωτές αυτό τον περιορισμό διότι μακροχρόνια Τη στιγμή που ε, επεκτείνεται η περιαγωγή μέσω διαδικτύου και βεβαίως ε, οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν υψηλό κέρδος για να υποστηρίξουν αυτές τις υπηρεσίες, τότε το roaming θα εξαφανιστεί, διότι στο διαδίκτυο θα είναι πολύ πιο φτηνό σε σχέση με τα κινητά. Δεύτερον, πολλοί συνάδελφοι ε, καταγράφω ότι θέλουν να υπάρχουν όρια τιμών ή ένα ε, σύστημα προειδοποίησης για τους ε, συνδρομητές όταν το τιμολόγιο τους υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο και αυτό αφορά όλες τις υπηρεσίες τηλεφωνίας. Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ότι ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών τιμών, ε, υψηλότερες ή χαμηλότερες και που σχετίζονται με την τιμολόγηση στις χώρες ε, των, ε, των πολιτών όπου στέλνουν SMS. Οι τιμές λοιπόν, η προσέγγιση αυτή μπορεί να γίνει αυθαίρετη τη στιγμή που μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα ε, υπηρεσιών που ε, παρέχει η υπηρεσία αυτή, μάλλον ο πάροχος διασυνοριακά. Και αυτό θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει και στην Επιτροπή και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυθαίρετα συμπεράσματα και μέτρα μιας βιομηχανίας που δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να το επιτύχουμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος οι αυθαίρετες τιμές ε, που προτείνονται. Άρα η Επιτροπή ας λάβει το λόγο και ίσως ε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και αυτά που αναφέραμε, δηλαδή την παρέμβαση στην αγορά που είναι ε, πολύπλοκη αγορά και ποιες εναλλακτικές διαγράφονται. Ίσως η βιομηχανία θα πρέπει να αυτορυθμιστεί και να μειώσει τις τιμές έτσι ώστε να μην χρειάζεται νομοθέτηση. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ήδη την ε, κατατελευταία σας συνεδρίαση είπα ότι η Επίτροπη εξετάζει αυτή την πρόταση σαν μια εξαιρετική περίπτωση. Αυτό κατέστη σαφές σε όλα μας τα έγγραφα στην ε, έκθεση αντικτύπου και όλες τις παρουσιάσεις της ε, Επιτροπής. Όπως ανέφερε και η Επίτροπος Ρέντινγκ παρακολουθήσατε τη συζήτηση με την έγκριση του πρώτου κανονισμού περί αγωγής. Γιατί δηλαδή αναλάβαμε δράση σε αυτή την αγορά. Έχουμε το νομικό πλαίσιο και διαθέτουμε και ένα σύστημα ανάλυσης της αγοράς με βάση το οποίο θα δούμε κατά πόσο υπάρχει ανταγωνισμός ή όχι και μετά κατά πόσο υπάρχει ρύθμιση. Η αγορά αναλύθηκε από πολλές εθνικές ρυθμιστικές αρχές και αφού συζήτησαν το ζήτημα, ζήτησαν να αναλάβει δράση η Επιτροπή γιατί δεν μπορούσαν μεμονωμένα να επιλύσουν το ζήτημα σε κάθε κράτος μέλος για την ρύθμιση της αγοράς σε ένα κράτος μέλος που θα επηρεάζει δυσμενώς ένα άλλο κράτος μέλος. Άρα ζήτησαν από την Επίτροπη να παρέμβει και να προτείνει έναν κανονισμό. Αυτό ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη φάση. Άρα η νομική βάση του κανονισμού είναι η εσωτερική αγορά και το πλαίσιο που μας απασχολεί σχετίζεται με την προστασία και του καταναλωτή. Με βάση αυτές τις αρχές φτάσαμε σε αυτόν τον κανονισμό και τώρα προτείνουμε αυτή την επέκταση. Και στην έκθεση αντικτύπου ε, βλέπουμε γιατί η αγορά μέχρι τώρα δεν ήταν λειτουργική. Όμως δεν προτείναμε αγορά ε, λιανικής με στοιχεία, διότι πολλοί είπατε στις ότι είναι μια αγορά η οποία κινείται εντάχει. Υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις και πιστεύουμε ότι ο κανονισμός περιχονδρικής αρκεί ως προς τις τιμολογήσεις και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει στην αγορά, δηλαδή ότι οι τιμές σε επίπεδο λιανικής δεν είναι τόσο υψηλές έτσι ώστε να πρέπει να δράσουμε σε επίπεδο λιανικής. Σε επίπεδο χονδρικής θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να δράσουμε διότι έτσι θα υπάρχουν οι κατάλληλοι όροι για τους ε, μικρότερους παρόχους έτσι ώστε να προβάλλουν προσφορές που να είναι ανταγωνιστικές στην αγορά. Η εργασία μας που σας ε, υποβάλαμε αφορά μια διαδικασία δημόσιας ε, διαβούλευσης με όλες τις αίρα και πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια λογική και αναλογική προσέγγιση. Επικεντρωθήκαμε σε θέματα διαφάνειας και μιλήσαμε για περικοπές. Όμως, πάροχοι μπορούν να, να προβάλλουν εναλλακτικέ λύσεις, άρα υπάρχουν οι περικοπές, αλλά οι πάροχοι μπορούν να προβάλλουν ε, μειώσεις ε, τιμών σε σχέση με τους καταναλωτές. Δηλαδή δεν μειώνουμε το φάσμα επιλογών, απλώς μπορεί να υπάρξουν ε, τέτοιες περικοπές έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό το σοκ τιμολογήσεων που αντιμετωπίσαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Επίσης πιστεύω ότι συζητήσαμε θέματα διαφάνειας και εκτάκτων μέτρων αλλά πιστεύουμε εν τέλει ότι αυτά που προτείνουμε βασίζονται στοιχεία και ιδιαίτερα στοιχεία κόστος που μας δίνει η βιομηχανία, δεν προσανατολιζόμαστε προς το κόστος, γιατί πιστεύουμε ότι η προσέγγιση του πρώτου κανονισμού θα πρέπει να ισχύει και στο δεύτερο, για να υπάρχει συνέπεια. Άρα επιτρέπουμε ένα περιθώριο κέρδους και κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι δώσαμε μια ευκαιρία στους παρόχους να αντιδράσουν. Η κυρία Ρέντινγκ ανέφερε επανειλημμένα και με επιστολές ότι αν δεν προτείνουν λύσεις θα πρέπει να τις προτείνουμε εμείς. Αυτό αφορά τους συνομοθέτες, τα τρία θεσμικά όργανα. Τα στοιχεία που έχουμε σήμερα δείχνουν ότι στο SMS υπάρχει σταθερότητα στα πλαίσια της ε, διεθνούς περιαγωγής ως προς το ε, φωνητικό roaming, τη φωνητική περιαγωγή. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στα όρια και ως προς την περιαγωγή δεδομένων κινούμαστε στην ε, σωστή κατεύθυνση ως προς τη χονδρική, αλλά έχουμε μικρά προβλήματα με τους μικρούς παρόχους. Ευχαριστώ. Ωραία λέει Πρόεδρος. Ο εισηγητής θα συνοψίσει. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα σημεία. Η κυρία Ρίς Γιόργενσεν είπε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμό στην αγορά περιαγωγής. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλοί πάροχοι που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες και μπορούμε να προστρέψουμε και σε άλλες υπηρεσίες. Και αν δούμε και τις διαθέσιμες τεχνολογίες, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν Wi-Fi και όχι ε, τα κινητά τους για τη μεταφορά δεδομένων. Και αυτό θα καταστρέψει την αγορά ε, περιαγωγής. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ρυθμίσουμε σήμερα για αύριο, γιατί μπορούμε να εξαφανίσουμε υπηρεσίες. Επίσης υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούν Αλλά υπάρχουν ε, και εκπτωτικές κάρτες σε σχέση με τη σχέση κόστους οφέλους θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση του κόστους και μιλάμε για τα κινητά ή για όλους τους τομείς. Εάν λάβουμε υπόψη μόνο τον τομέα της κινητής, αν δείτε την τιμολόγηση των συσκευών, αν θέλουμε να κινηθούμε προς το κόστος, τότε θα πρέπει να πούμε σε όλους τους πελάτες ότι θα πρέπει να καταβάλουν και ένα ε, μέρισμα του κόστους της συσκευής αντί να μην καταβάλουν τίποτα ή ένα πολύ ε, μικρό αντίτιμο. Σε σχέση με το Sunset Regulation, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Και ως προς το σοκ της τιμολόγησης υπάρχει συμφωνία σε αυτή την Επιτροπή ότι χρειάζεται διαφάνεια. Και αυτό που προσπάθησα να κάνω στις τροπολογίες μου είναι να λάβει πληροφορίες ο καταναλωτής όταν μπαίνει στην αγορά, όταν κάνει περιαγωγή, όταν κάνει λόγκον, όταν έχει διασυνοριακές συναλλαγές. Στις τροπολογίες μου Προτείνω, αντί να έχουμε ad hoc μέτρα διαφάνειας, να έχουμε συνεκτικά και εκτενή μέτρα. Και αυτό το γνωρίζουν αυτοί που συνεργάζονται με πάροχους κινητής τη στιγμή που προτείνουν νέα πακέτα στους καταναλωτές. Δηλαδή, ως προς την τιμολόγηση, τα στοιχεία τιμολόγησης έρχονται πολύ αργά. Δηλαδή το τμήμα τιμολόγησης αργεί πάρα πολύ. Άρα μπορούμε να, δώσουμε, να έχουμε μια μεγαλύτερη πλαισίωση για όλα ή να ζητήσουμε την σταδιακή εισδοχή της ε, υπηρεσίας ε, τιμολόγησης. Ως προς τα προπληρωμένα, τις προπληρωμένες κάρτες, εδώ χρειάζεται μία νέα αναβάθμιση και προσαρμογή, αλλά θα πρέπει να δώσουμε στον καταναλωτή όλο ένα και περισσότερες πληροφορίες στο συνάδελφο Χάνσλετ. Δεν ξέρω κατά πόσο η ρύθμιση τιμών θα οδηγήσει σε περισσότερο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα προς, ως προς τους μικρούς ε, παρόχους, γιατί πολλοί ε, καθαροί εισαγωγείς ανησυχούν για το μέλλον τους γιατί υπάρχουν στην χώρια αγορά αλλά πουθενά αλλού και δεν ξέρουν τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στα έσοδα τους τη στιγμή που ίσως να μην μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν στην αγορά. Σε μία ε, μικρή χώρα μου είπε ένας τέτοιος ε, εισαγωγέας ότι θα κάνει μικρές επενδύσεις στη χώρα του και μεγάλες επενδύσεις ε, διασυνοριακά. Άλλοι μου είπαν ότι θα περιορίσουν τους ε, καταναλωτές, τους πελάτες και είπαν ότι δεν μπορούν να επεκταθούν στην περιαγωγή, αλλά στις ε, τιμές προτείνεται δεν υπάρχει καμία οικονομική βάση. Ο Μάλκομ Χάρμπορ είπε ότι είναι αυθαίρετες οι τιμές, αυθαίρετη η τιμολόγηση. Κύριε Σμίτ, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Αν ε, διαβάσετε το βιβλίο The Road to Serfdom, Βλέπετε ότι όλοι, θέλουν, όλοι που θέλουν κρατικό παρεμβατισμό θεωρούν ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για υπέρ των καταναλωτών, υπέρ των μικρών παρόχων, ότι το κέρδος είναι πολύ κακό και θα πρέπει να υπάρχει δημόσια και κρατική παρέμβαση, καθώς και κρατισμός. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Συμφωνώ με τον κύριο Χάρμπορ για τις αυθαίρετες τιμές και θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί στον ανταγωνισμό. Στην κυρία Μισού από την Επιτροπή, ξέρω ότι είπατε ότι είναι προσωρινό το μέτρο και ε, εξαιρετικό, δηλαδή έκτακτο, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν υπήρξε ε, η φορολόγηση του εισοδήματος αρχικά ήταν προσωρινό το μέτρο, αλλά ισχύει. Ο Μίλτον Φρίντμαν είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μόνιμο από ένα προσωρινό κυβερνητικό σχέδιο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία λοιπόν από τους πάντες. Συνένεση λοιπόν. Θα ψηφίσουμε. 2 Μαρτίου, 2 Μαρτίου, έτσι δεν είναι, κύριε Σιγητά. Ωραία. Άρα έχετε χρόνο να το συζητήσετε, εάν συμφωνείτε. Διαφορετικά θα δούμε ποια πλειοψηφία θα κερδίσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Καμάλ, τον εισηγητή μας και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα έτσι ώστε να αποχωρήσουν όσοι το επιθυμούν. Η έκθεση Μάντερς λοιπόν είναι το επόμενο θέμα. Κύριε Μάντερς, έχετε το λόγο. Ο κύριος Μάντερς είναι εδώ. Και θα μιλήσουμε για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως ανηλίκων, όσο αφορά τη χρήση, βίντεο παιχνιδιών. Έχουν υποβληθεί τροπολογίες 14 νομίζω, άρα όχι και πολλές. Άρα θα φτάσουμε σε συμφωνία σε επίπεδο επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον εισηγητή μας να μας παρουσιάσει το σχέδιο ε, γνωμοδότησης και να μας μιλήσει και για τις τροπολογίες. Μάντερς. Ευχαριστώ. Μπορεί να είμαι σύντομος διότι Υπάρχει ευρύτατη συνένεση στο Κοινοβούλιο, 14 μονοτροπολογίε έχουν κατατεθεί, συνένεση τουλάχιστον σε ό,τι φορά τα βίντεο παιχνίδια συνένεση έλεγα για το ότι τα βίντεο παιχνίδια, επαναλαμβάνω, έχουν θετικές ε, επιπτώσεις στις κοινωνίες μας. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες απειλές, αλλά αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα. Αν φάει κανείς πολλές πίτσες δεν θα το κάνει καλό. Εξαρτάται λοιπόν πώς ε, χρησιμοποιείται το παιχνίδι και την πίτσα. Επίσης ε, το σύστημα PEGI λειτουργεί ικανοποιητικά, πως υπάρχει ένα σύστημα ε, υπολογισμού, ε, διαβάθμισης και, τα... και μπορεί φυσικά να βελτιωθεί περαιτέρω. Θεωρούμε ότι το σύστημα PEGI μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των γονιών αλλά και των δασκάλων διότι πολλές φορές βλέπουμε ηλικιωμένα άτομα όπως εγώ να μην αρέσκονται σε καινοτομίε, σε νεοτερισμού κλπ. Αλλά είναι, και είναι επίσης δύσκολο να τα συνηθίσουν, να εξοικειωθούν. Αλλά τα παιδιά μου όμως παίζουν με βίντεο παιχνίδια, ενώ εγώ όχι. Το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά συστήματα για την ηλικιακή διαβάθμιση και πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να αποκτήσουμε ένα σύστημα διαβάθμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γνωμοδοτήσεις των συναδέλφων στην Επιτροπή Πολιτισμού και ΛΥΜΠΕ ε, κάνουν κάποιες ε, συστάσεις ε, τις οποίες μπορώ να δεχθώ. Υπάρχουν ορισμένες τουλάχιστον δύο επί των οποίων θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια συμβαστική λύση και να τονίσω πως γενικά Συμφωνούμε επί του θέματος να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους για την συνεργασία και για τις προτάσεις, για την στήριξη που μου δώσανε, αλλά και τη γραμματεία. Και πιστεύω πως η τελική ψηφοφορία θα οδηγήσει σε μια βελτίωση της αντιμετώπιση των βίντεο παιχνιδιών και όπως είπε ο καθηγητής Goldsmith, αυτό θα αποτελέσει για μια στήριξη της ε, του κοινωνίες μας και του μέλλοντος μα, Κύριε Σαγγέλακας. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι και εγώ σύντομο. Ε, τα βιντεοπαιχνίδια είναι δημοφιλή, πολύ δημοφιλή μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων στην Ευρώπη με μια αξιοσημείωτη αγορά πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Τα βιντεοπαιχνίδια είναι χρήσιμα διότι βοηθούν τους νέους να οξύνουν την κρίση τους, την αντίληψή τους αλλά κρύβουν και κινδύνους και αυτό ακριβώς προσπαθούμε εδώ να μελετήσουμε και πρέπει να πω ότι ο εισηγητής μας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην προσπάθεια να περιγράψει τα προβλήματα και τους κινδύνους. Ε, νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα συμβάλλει, θα δώσει ένα κίνητρο παραπέρα στην ε, οριοθέτηση και τους τρόπους λειτουργίας των ε, Έχω καταθέσει ορισμένες ε, τροπολογίες που περισσότερο σχετίζονται με την ανάπτυξη των συστημάτων PEGI και PEGI Online, με την ευαισθητοποίηση των γονέων και κηδεμόνων να ασχολούνται και να παρακολουθούν πού βρίσκονται τα παιδιά τους όταν, και με τι ασχολούνται όταν ασχολούνται με τα βίντεο παιχνίδια, με, τον, με τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να πάρουν τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε τουλάχιστον σε κάποια κράτη-μέλη όπου βιντεοπαιχνίδια βρίσκονται σε ίντερνετ καφέ, να υπάρχει μία οριοθέτηση ε, πάνω στο τι, με τι ασχολούνται τα παιδιά, πόσες ώρες ασχολούνται και με το περιεχόμενο των βίντεο παιχνιδιών και επίσης με ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργάζονται με μια άλλη τροπολογία στενά όσον αφορά την προώθηση της προστασίας των ανηλίκων. Κλείοντας να πω ότι τα βιντεοπαιχνίδια είναι χρήσιμα, μέχρι και στην ιατρική έχουν εφαρμογές, αλλά ταυτόχρονα κρύβουν κινδύνους για τους οποίους όσοι εδώ σε αυτή την αίθουσα είναι γονείς, καλό είναι να ανησυχούν και να είναι προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Okay. Uh, have I got any other members that want to intervene? I think most people are happy with the approach that the rapporteur has taken, and I think. Νομίζω ότι μια που υπάρχουν λίγες ε, τροπολογίες, υπάρχει κατά μάλλον το συνένεση, υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω πως η προσέγγιση του Κοινοβουλίου επί του θέματος συμπίπτει κατά ένα σημαντικό βαθμό με αυτήν της Κομισιόν. Η ενημέρωση των γονέων έχει τεράστια σημασία. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω πως υπάρχουν περαιτέρω σχόλια. Έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις της ε, πολιτισμού και ΛΥΜΠΕ. Επανέρχομαι στον εισηγητή. Από ό,τι φαίνεται είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχουν ε, διαφορές. Κύριε Μάντερς. Ναι, φυσικά και μπορούμε να ψηφίσουμε. Και ελπίζω πως ε, θα βελτιώσουμε την ε, κατάσταση. Όπως είπε και η Κομισιόν θα πρέπει να ενημερωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι γονείς και το σύστημα ΠΕΓΙ e μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν υπάρξουν παράπονα από τους γονείς ε, το σύστημα ΠΕΓΙ μπορεί να λειτουργήσει και ελπίζουμε λοιπόν στο μέλλον, το μέλλον ακόμα και οι γονείς που δεν γνωρίζουν πολλά περί ε, υπολογιστών και διαδικτύου να μπορούν να πατούν ένα κουμπί για να απαγορεύουν κάποια προγράμμα, παιχνίδια. Κομισιόν, έχει να πει κάτι, όχι. Πρόκειται για ανακοίνωση δεν απαιτείται περί νομοθεσία περί του θέματος, αλλά να υπάρξει το δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία. Τι όρθιο ψηφίσουμε αύριο. Μήπω θα πρέπει να φέρετε και τις κάρτες σα αύριο, επειδή υπάρχουν πολλέ τροπολογίε. Καλό να έχετε τις κάρτες. <coughs> Καλού κακού. Για να είμαστε ταχύτεροι. Ή άμα οι ψηφοφορίες ε, έχουν κάποιο πρόβλημα, ε, ε, δεν είναι σαφής η αμα οι ψηφοφοριε εχουν καποιο προβλημα δεν ειναι σαφης η πλειοψηφια αν υπάρχει διαφορά στήθους. Εντάξει, θα στείλουμε ένα mail στους συναδέλφους αν δεν τις φέρετε μπορεί να χρειαστείτε να πάνε τις πάρετε. Ένα πεντάλεπτο χρειάζεστε. Εντάξει, ολοκληρώσαμε. Αύριο στις ψηφοφορίες θα τα πούμε. Γεια σας.